Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κηρύσω εδώ την ε, συνέχιση της ε, συνεδρίασης της Συνόδου Ολομελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεκόπη την 5η 19 Φεβρουαρίου του 2009. Αγαπητοί συνάδελφοι και ομιλώ στην γλώσσα της χώρας η οποία επλήγει από το φοβερό αυτό περιστατικό. Θα μάθατε μάλλον τα λυπηρά γεγονότα της επιθέσεως του Σαββατοκύριακο στην Βόρεια Ιρλανδία εναντίον μιας Βρετανικής βάσης που ε, κόστη τη ζωή σε δύο